παρεμβάσεις και έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Το περνάμε το ψήφισμα από τέσσερις ε, ομάδες. Περνάμε τώρα στην υπόθεση του Ελ Σαλβαδόρ και των γυναικών που διώκονται. Ο κύριος Γιούρεκ. Γιούρεκ Μάρεκ, ο Ελ Σαλβαδόρ ε, είναι ένα, ένα δημοκρατικό καθεστώς, μια δημοκρατική χώρα που θέλει να προστατεύσει τη ζωή. Και μάλιστα και το Freedom House και το Economist το έχει ψηλά σε αυτή τη λίστα. Και παρόλα αυτά δέχεται επι, ε, επιθέσεις επειδή θέλει να προστατεύσει τη ζωή. Ακόμη και απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται τέτοιες επιθέσεις. Θα πρέπει να σταματήσουμε να θέτουμε όρους και να συζητήσουμε για τεχνικούς τρόπους πώς θα μπορούμε να προσπίσουμε το δικαίωμα στη ζωή. Γιατί μόνο αν συμφωνήσουμε γι' αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε πώς θα το προσπίσουμε. Διαφορετικά υπερασπίζουν το δικαίωμα στη ζωή η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, το Ερ Σαλβαδόρ. Αυτό το δικαίωμα προϋποθέτει μια ενίσχυση των ε, κανόνων Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σίγουρα η Πολωνία είναι από πιο ασφαλείς χώρες στην οποία γίνεται σεβαστή η ζωή. Ε, το Ελ Σαλβαδόρ ε, νομίζω ότι δεν είναι ε, ένοχο, γιατί είναι η μόνη χώρα που πραγματικά προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν καταπατά. Σας ευχαριστώ. Σκοτ Κέιτο για ένα λεπτό. Με ναι, μικρόφωνο παρακαλώ. τον Σεπτέμβριο επισκέφθηκα την φυλακή Ιλαπάγκα κατά την διάρκεια της επίσκεψης της αποστολής μας. Σοκαρίστηκα. Οι γυναίκες είχαν φυλακιστεί λόγω του ότι είχαν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και σε κάποιες περιπτώσεις λόγω αποβολής ή βιασμού. Είναι μεγάλο πρόβλημα η βία με βάση το φύλλο στο Ελσαλβαδόρο που έχουμε συχνά διασμούς και αιμομιξίες που καταλήγουν σαν της εγκυμοσύνης από το 1998 έχει απαγορευτεί η έκτρωση σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και όταν απειλείται η ζωή της εγκύου ή όταν δεν είναι βιώσιμο το έμβριο. 14 γυναίκες πέθαναν ε, πέρσι ε, από επιπλοκές που είχαν σχέση με την έκτρωση. Γνωρίζουμε πως το Ελσαλβαδόρ προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση και αναγνωρίζουμε το έργο των Ευρωπαίων διπλωματών. Ελπίζουμε το ψήφισμα αυτό να ευστήσει την προσοχή όλων ε, στα προβλήματα γυναικών ε, όπως η Μπεατρίς ε, Δεκρούς οι οποίες θα έπρεπε να έχουν λάβει χάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σουρμπάν Κρέσπο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ διεκδικούμε την ελευθερία της Βάσκες, της Εμελίνα Αρμάντες και όλων των γυναικών που έχουν φυλακιστεί στο Ελσαλβαδόρ είτε επειδή απέβαλαν είτε επειδή υπέστησαν ανεπιθύμητες ε, εκτρώσεις. Θέλουμε αποποινικοποίηση τη έκτρωση όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε όλε τι υπόλοιπε που απαγορεύουν την άβλωση ή που την επιτρέπουν μόνο υπό συγκεκριμένου όρου γιατί ε, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι δικαίωμα των γυναικών και γι' αυτό θα πρέπει η διακοπή της εγκυμοσύνης να γίνεται με ασφαλή τρόπο. Οι δεμοί παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και αξιοπρέπειά τους. Και η ισότητα των δύο φύλων δεν πρόκειται να ε, γίνει ε, πραγματική αν δεν εξασφαλίσουμε την ελεύθερη απόφαση των γυναικών για το σώμα τους και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσουν για την ασφαλή και ε, ξεκάθαρη πρόσβαση όλων των γυναικών στην αποβολή. Όχι μόνο στο Ελσαλβαδόρ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Πρέπει να εγγυηθούμε αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρουμπάν Κρέσπο. Το λόγο η κυρία Μπεσέρα Μπαστερετσέα. Στο Ελσαβαδόρ η έκτρωση απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά από βιασμό. Και μάλιστα ε, επισύρει ποινή μέχρι και 30 ετών κάθερξη, όπως τα κακουργήματα στην Ευρώπη. Ε, ακόμη και σε περίπτωση αυθόρμητης αποβολής, ε, ε, η κυρία Χερνάντες ε, ήταν θύμα βιασμού, είχε θνησιγένεια και παρόλα αυτά βρίσκεται στις φυλακές με ποινή φυλάκισης, όπως η Θεοδόρα Δεκάρμεν Μπάσκες, που η ποινή της επιβεβαιώθηκε από το δικαστή και άλλες γυναίκες. Είναι πραγματικά απαράδεκτη και ασυνήθιστη αυτή η εις βάρος των γυναικών σε μια χώρα που είναι από τις πιο βίες της περιοχής και του κόσμου. Πρόκειται για μια τιμωρία που την επιβάλλουμε ακόμη και σε θύματα, σε θύματα βιασμού. Ουσιαστικά η χώρα αυτή μπλοκάρει την ανάπτυξη, την εξέλιξή του και δεν μιλούμε μόνο για την ελευθερία. Η ποινικοποίηση Τη έκτρωσης ε, βάλει κατά της ίδιας της υγείας ε, και της ελευθερίας των γυναικών και λυπάμαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη βούληση και δεν έχει καταλήξει συνένεση για να ζητήσουμε αποποινικοποίηση της ε, έκτρωσης σε κάθε περίπτωση και δυνατότητα έκτρωσης υπό όρους έστω σε μερικές περιπτώσεις στο Σαλβαδόρο Αποζήτησαν και τα Ηνωμένα Έθνη ο ειδικός εντεταλμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπεσέρα Μπαστερετσέα. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σωράγια Πόστ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τις αρχές του Σαλβαδόρ, ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε για τη ζωή, για το σώμα των γυναικών. Πώς μπορείτε να καθαριστάτε ποινικό αδίκημα την αποβολή εμείς εδώ οι ευρωβουλευτές με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα υψώνουμε το ανάστημα έναντι των παραβιάσεων των δικών σας. Τα κράτη και οι εκκλησίες δεν έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας. Το σώμα μου είναι το σώμα μου και είναι δική μου απόφαση εάν θα κάνω αμβλώση ή όχι. Κάθε γυναίκα στον κόσμο έχει το δικαίωμα να προβεί σε αυτή την επιλογή για τον εαυτό της. Υψώνουμε το ανάστημα για να στηρίξουμε τις γυναίκες που έχουν ε, πέσει θύματα αυτών των νόμων. Να απολευθερωθούν λοιπόν οι γυναίκες από τη φυλακή, από τις αρχές του Σαλβαδόρ και να καταργηθούν οι νόμοι που υποχρεώνουν τα νοσοκομεία να καταγγέλουν όποια γυναίκα έρχεται να ζητήσει την ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην αστυνομία πρέπει να ε, αγωνιστούμε για κάθε για να καταργηθεί κάθε μορφή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και ως γυναίκα και ως πολιτικός Ψήνω το ένα μου και στέκομαι δίπλα σε κάθε γυναίκα και στο δικαίωμά της να αποφασίζει για τη ζωή της. Σήμερα ακούσαμε τα νέα της Θεοντόρα Μπάσκες ότι δηλαδή η α, έφεση τη ε, απερίφθη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται η καταδίκη της σε 30 χρόνια φυλάκιση. Αυτό είναι ντροπή για το Ελσαρβαδόρ. Κύριε Γιούρε, και εσείς το βρίσκετε σωστό 30 χρόνια να μείνει καταδίκη στην φυλακή. Είναι δυνατόν να κοιτάτε οποιοδήποτε άνθρωπο στα μάτια. Ντροπή σας. Καλώς ευχαριστώ. Και έχετε μία μπλε κάρτα, κυρία Πόστ. Δέχεστε την ε, ερώτηση με μπλε κάρτα του κυρίου Λούτκε. Λούκε. Τη δέχεστε την κάρτα του κυρίου Λούκε. Όχι κύριε Λούκε. Η κυρία Απόστη δεν δέχεται. Ε, έχω δικαίωμα να απαντήσω. No Καλώς, λοιπόν, προχωρούμε. Κατάλογος των ε, ομιλητών. Απερίφθη το αίτημα για μπλε κάρτα του κυρίου Λούκε, λέει η ομιλήτρια. Η κυρία Κοσλός, Κοσλόφσκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μιλούμε για το Ελ Σαλβαδόρ, μια μικρή χώρα στην Κεντρική Αμερική, που πρόσφατα το 1998 απαγορεύθηκε πλήρως το δικαίωμα στην έκτρωση. Ακόμη και η γυναίκα που έχει υποστεί βιασμό και έχει εγκυμοσύνη που απειλεί τη ζωή της δεν μπορεί να κάνει άμβλωση. Αυτό είναι απαράδεκτο και μάλιστα στο Ελσαλβαδόρ ο νόμος ερμηνεύεται με τρόπο που αρνείται τις, ε, τα επιστημονικά πορίσματα, ακόμη και το τεκμήριο της αθότητας. και γυναίκες αβάσιμα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, για παιδοκτονία ή για εσκεμμένη διακοπή της δικαιοσύνης και φυλακίζονται για πολλά, της εγκυμοσύνης και ε, φυλακίζονται για πολλά χρόνια. Ε, μάλιστα πολλές φορές ε, ανήλικα κορίτσια ε, έγκυες ε, διαπράττουν αυτοκτονία. Οι ποινές είναι ποινές κάθυρσης, κάθυρξης πολλών χρόνων και μάλιστα οποιαδήποτε αποβολή, ακόμη και είναι αυθόρμητη, δημιουργεί υπόνοιες για εσκεμμένη διακοπή της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό και μερικές φορές ε, οι γυναίκες αποφεύγουν ε, να προσφύγουν στα νοσοκομεία ή σε γιατρούς γιατί τις καταγγέλουν. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε το Ελσαλβαδόρ να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και να αποφυλακίσει αυτέ τι γυναίκε, στηρώντα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι αδύνατον τέτοια δικαιώματα όπω το θεμελιώδη δικαίωμα στην ε, ελευθερία να ε, τιμωρείται ποινικά. Άλλωστε, κύριε Γιούρεκ, ε, το πολωνικό δίκαιο δεν έχει καμία σχέση με το δίκαιο που ισχύει στο Ελσαλβαδόρ. Και μάλιστα στην μαύρη πορεία 100.000 γυναίκες κατέβηκαν στην, στους δρόμους στην Πολωνία διαδηλώνοντας κατά της ε, απαγόρευσης ε, του δικαιώματος έκτρωσης. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τις γυναίκες αυτές. Ο κύριος Γιούρεκ έχει ζητήσει μια μπλε κάρτα. Κυρία Κοσλόφ Σκαράιεβιτς, δέχεστε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ακούσατε πριν πριν από λίγο ότι ε, το, το έμβριο είναι τμήμα της, ε, του σώματος της γυναίκας. Ε, πιστεύω ακριβώς ότι γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά του. Και αυτό προβλέπει και το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Πολωνία. Γιατί είστε κατά της προστασίας της ζωής, του δικαιώματος στη ζωή. Η κυρία Κοζουόφσκα Ραϊέβιτς. Κύριε Γιούρεκ, το πολωνικό δίκαιο ε, περιλαμβάνει τρεις εξαιρέσεις από την απαγόρευση της ε, έκτρωσης. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο Ελσαλβαδόρ. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε συντηρητικό δίκαιο που παρόλα αυτά προστατεύει η ζωή και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα της γυναίκας ως ε, πλήρους πολίτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στους ομιλητές ε, εξ των πολιτικών ομάδων. Για τους σοσιαλδημοκράτες, ο Φρανσίσκο Ασής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Τεοντόρα Βάσκες εδώ και δέκα χρόνια είναι φυλακισμένη και έχει ε, της έχει επιδικαστεί 30 ετής ε, ε, ποινή για ποιο έγκλημα επειδή γέννησε νεκρό έμβριο. Και είναι και άλλες γυναίκες σε αυτήν την κατάσταση. Το παρόν ψηφίσμα υιοθετεί μια ηχηρή πολιτική θέση για την περίπτωση της Θεοδόρας και άλλων γυναικών που υπέστησαν την ίδια βαναυσότητα, ιδίως την ομάδα των 17 γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή εκτίοντας ποινές δεκαετιών Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να ασκήσει πιέσει στις ε, αρχές του Σαλβαδόρ για να ανατρέψουμε αυτή την άδικη κατάσταση για τις γυναίκες. Γιατί ε, θα πρέπει επιτέλους να γίνει δημόσια συζήτηση στο Ελσαλβαδόρ για την αποποινικοποίηση της έκτρωσης. Είναι πραγματικά πολύ τολμηρές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που προωθούν και νομίζω ότι υπάρχει και μια νομοθετική πρόταση για μια έκτρωση πιο αξιοπρεπή και πιο ανθρωπιστική. Θα ήθελα να ενθαρρύνουμε το Ελσαλβαδόρ για να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση και να σταματήσει αυτό το βάναυσο και απάνθρωπο θέμα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη χώρα. ευχαριστώ πάρα πολύ. μιλήνα για ένα λεπτό. Κύρια Πρόεδρε, οι συντηρητικές δυνάμεις στο Ελσαλβαδόρ θεωρούν τις γυναίκες και τα παιδιά μόνο ως μηχανές αναπαραγωγής. Και βλέπουμε ότι βλέπονται ποινές φυλάξεις μέχρι 8 χρόνια για τις αποβολές και μέχρι και 50 χρόνια για τις εκτρώσεις. Δηλαδή αυτά ακούγονται σαν εφιάλτης, αλλά είναι καθημερινή πραγματικότητα για τις γυναίκες και τα παιδιά στο Ελσαλβαδόρ εν 2017. Για όσους από εμά εδώ μέσα θεωρούμε ότι αυτά δεν είναι δουλειά μας και ότι σώζει ζωές, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσες γυναίκες και παιδιά πρέπει να υποφέρουν μέχρι να καταλάβετε ότι είναι κοινικό αυτό. Σκοτώνετε ανθρώπους και υπερασπίζετε τον φόνο. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως δεν θα εγκαταλείψω αυτά τα, αυτές γυναίκες και τα κορίτσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ράιντ και για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Θεοδόρα και η Εύελεν είναι δύο γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει φοβερά πράγματα στη ζωή τους. Όχι μόνο είχαν αποβολή, αλλά τώρα κατηγορούνται και για φόνο και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης. Πολυετή. Προς τις αρχές του Σαλβαδόρ απελευθερώστε την Θεοδόρα, την Εύελιν και όλες τις άλλες γυναίκες που έχουν φυλακιστεί για αποβολή. Ο νόμος του Ελ Σαλβαδόρ είναι η νομοθέτηση του μισογενισμού. Πρόκειται για μια αναζήτηση της απόλυτης κυριαρχίας της πατριαρχίας επί του σώματος των γυναικών. Το σώμα τους ανήκει στις ίδιες και όχι στο κράτος. Οι γυναίκες έχουν και αυτές δικαίωμα στη ζωή. Δικό μου το σώμα, δικά μου τα δικαιώματα. Ε, Ευχαριστώ πολύ, <coughs> Κύριε Ράντκε. Η κυρία Γκαρσία Πέρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Θεοδόρα Δε Κάρμερ είναι 34 ετών και πάνω από 10 χρόνια βρίσκεται στις, φυ στις φυλακές. Στις φυλακές επειδή έχασε σε, μια πρόορη, σε ένα πρόωρο την κόρη της και χθε οι αρχές του Ελσαλβαδόρ επιβεβαίωσαν την 30 της κάθερξη. Ποινικοποιείται το, η αποβολή ε, ε, κρίνονται ένοχε οι γυναίκες του Σαλβαδόρα ακόμη και σε περίπτωση αυθόρμητες αποβολής. Ε, και μάλιστα ε, βρίσκονται στις φυλακές και μαραζώνουν με στερητικές τις ελευθερίες ποινές. Σε πολλές περιοχές του κόσμου στερούμε τη, την ελευθερία των γυναικών και το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για τη ζωή τους. Θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερική πολιτική και η πολιτική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εγγυώνται τα δικαιώματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας όλων των γυναικών του κόσμου. Γιατί ο δικός τους αγώνας είναι και δικός μας αγώνας. Το σώμα μας είναι η ελευθερία και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας στην Ευρώπη για να έχουν πρόσβαση στην ελευθερία όλες οι γυναίκες του κόσμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαρσία Πέρες. Το λόγο έχει τώρα με τη διαδικασία του Catch the Eye ο κύριος Πόλτσακ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν ο κύριος ε, Γιούρεκ ε, ε, εκφώνησε την ομιλία του, νόμιζε ότι μιλούσε για άλλο θέμα. Ούτε κουβέντα για την αλληλεγγύη προς τις γυναίκες, γυναίκες που είτε λόγω θνησιγένειας είτε λόγω αυθόρμητης αποβολής καταδικάζονται σε φυλάκιση. Δεν είμαι εγώ υπέρ των εκτρώσεων ιδιαίτερος, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες συνθήκες, κάποιοι όροι. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την ελεγγύη μου προς τις γυναίκες αυτές στο Ελ Σαλβαδόρ που έχουν πληγεί από τη σχετική νομοθεσία και έχουν φυλακιστεί μόνο και μόνο επειδή έχουν αποβάλει. Θα πρέπει να καταδικάσουμε αυτή την απαράδεκτη νομοθεσία όλοι οι λογικοί άνθρωποι, ακόμη και οι εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Γιούρεκ έχει ζητήσει μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Μάλιστα. Όχι. Καλώ προχωρούμε. Ο κύριο Καπούτο είναι ο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συζήτηση για την άμβλωση πάντοτε γυρεί ερωτήματα που μας φέρουν ενώπιον των συνειδήσεών μας πολιτιστικά και θρησκευτικά ζητήματα γύρονται και λαμβάνονται διαφορετικέ επιλογέ σε όλο τον κόσμο. υπάρχει μία κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί ποτέ να ε, ξεπεράσει κανεί τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια τη γυναίκα. Δηλαδή, ενώ το Ελ Σαλβαδόρ είναι το πιο καταπιεστικό προ τα δικαιώματα των γυναικών κράτο. Ένα από τα πιο καταπιεστικά. Η Μπεατρή Θερνάρντε Κρού έχει καταδικαστεί σε 30 ε, χρόνια φυλάκιση λόγω αυτόματης αποβολής εγκυμοσύνης, μάλιστα η οποία είχε προκληθεί από βιασμό. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε το σεβασμό της ε, γενετήσης αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων της γυναίκας. Μεταξύ αυτών είναι και η ασφαλής αποβολή. Εάν αυτό δεν επιτρέπεται, η ασφαλής άμβλωση καλύτερα. Εάν αυτό δεν εξασφαλιστεί, έχουμε να κάνουμε σοβαρότατη παραβίαση των δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν οι αρχές να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να αποφυλακιστούν οι γυναίκες οι οποίες είτε άθελά τους είτε σκεμμένα με άμβλωση έχουν αποβάλει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπούτο. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο Σαλβαδόρ συμβαίνει κάτι το απίθανο η νομοθεσία επιβάλλει ποινή φυλάκισης σε περίπτωση που γεννηθεί νεκρό ένα έμβριο ή συμβεί αποβολή. αυτό είναι το κεντρικό θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλες οι πλευρές αυτής της αίθουσας το καταγγέλνουν διότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και δεν είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι κάθε έμβριο το οποίο γεννιέται νεκρό ή σε περίπτωση πρόωρης αποβολής υπάρχει ευθύνη της μητέρας και αυτή να οδηγείται στις φυλακές. Κραυγαλαία περίπτωση είναι αυτή της Εύελιν η οποία έχει καταδικαστεί σε 30 χρόνια φυλάκιση και της αποδίδεται ανθρωποκτονία. νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά τα κεντρικά ζητήματα πρέπει να επικεντρωθούμε διότι αυτό είναι μια πρακτική στο σαλβαδόρ καθώς έχουν καταδικαστεί πάνω από 147 τουλάχιστον γυναίκες. αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αυτό το κεντρικό σημείο υπάρχει ενότητα νομίζω όλων των πλευρών εδώ και είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταδικάσουμε. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαριά. Ερνέστ Ουρτασούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από το 1998 ε, η έκτρωση απαγορεύεται και μέχρι το 2000 ε, χιλιάδες γυναίκες έχουν διωχθεί, έχουν ε, καταδικαστεί μέχρι και σε 30 χρόνια Σκεφτόμαστε σήμερα την Θεοδόρα που ήδη έχει συμπληρώσει 10 χρόνια στη φυλακή, η Εύελιν 18 ε, χρόνια και έχει άλλα, είναι 18 χρόνια και έχει άλλα 30 χρόνια να εκτίσει την ποινή της στη φυλακή. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε την ελευθερία αυτών των γυναικών και να γίνουν νομοθετικές αλλαγές για να ε, τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο του Σαλβαδόρ υπάρχουν κάποιε νομοθετικέ πρωτοβουλίε για τη μεταρρύθμιση του νόμου. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια όθηση σε αυτέ τι νομοθετικέ αλλαγέ για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Η αντιπροσωπεία μα του Ελ Σελβαδόρ κάνει πολύ καλή προσπάθεια από αυτή την άποψη και είναι πολύ σημαντικό εν ώψη των εκλογών του επόμενου έτου να συμβάλλουμε σε μια ουσιαστική και ρηξικέλευθη αλλαγή για να αποφυλακιστούν αυτέ οι γυναίκε, να απελευθερωθούν και ποτέ στο μέλλον να μην διώκεται μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή έκανε έκτρωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Ουρτασούν. Τώρα έχουμε έναν που έχει ζητήσει τον λόγο συγκεκριμένο. ο κύριο Καν, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, από το 1998 οι εκτρώσεις ποινικοποιούνται στο Ελσαλβαδόρ υπό οποιασδήποτε συνδίκη, οποιαδήποτε είναι καηφίσατε την υποψία έκτρωσης, ακόμα και στην περίπτωση αποβολής κινδυνεύει να φυλακιστεί. Πολλές έχουν φυλακιστεί και πολλές έχουν πεθάνει λόγω επιπλοκών. Πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος ε, προκαλεί μόνο πόνο σε γυναίκες ε, και στις οικογένειές τους. Και ακούσαμε χθες ότι το ίδιο θα γίνει και με την κυρία Βάσκες. Πρόκειται για ένα ε, δείγμα οπισθοχώρησης για τα δικαιώματα των ε, γυναικών. Πρόκειται λοιπόν για παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Ζητάμε από το Κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ να μεταρρυθμίσει τον ποινικό κώδικα και να αποποινικοποιήσει την έκτρωση υπό ορισμένες συνθήκες. Επίσης, να περάσει ένα μορατόριο στην εφαρμογή του ισχύοντος νόμου. Στις γυναίκε του Ελσαλαδόρ λέμε δεν είστε μόνες, είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Καν. Ε, για διαδικαστικό ζήτησε το λόγο ο κύριος Γιούρεκ. Θα ήθελα να επικαλεστώ το άρθρο 164 του εσωτερικού κανονισμού και σε περίπτωση προσωπικής αντέκλησης να μου δώσετε το δικαίωμα να απαντήσω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή και της κυρίας Πόστ ε, και του κυρίου Πόλτσακ ότι συνέχεια ε, μιλάτε για κάποια στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας. Μιλούμε για μια οργάνωση που και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επανειλημμένως ε, Αυτό παρουσιάστηκε ως ε, οργάνωση που είναι υπέρ της έκτρωσης, που δεν αντιμετωπίζει το έμβριο ως ανθρώπινο πλάσμα, αλλά ως κύμα που μπορεί η γυναίκα ελεύθερα να αποφασίσει να, να κάνει ε, έκτρωση ή όχι. Μην επικαλείστε λοιπόν τέτοιου είδους μονομερείς διεθνείς οργανώσεις για να στηρίξετε τα επιχειρήματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Βέλα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει βεβαίως ε, το τι συμβαίνει. Δεν ε, σχολιάζουμε αποφάσεις δικαστηρίων, αλλά σημειώνουμε με ανησυχία ότι σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλονται οι μέγιστες προβλεπόμενες ποινέ για γυναίκες οι οποίες απέβαλαν στο Ελ Σαλβαδόρ. Ο σεβασμός για το κράτο δικαίου είναι θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στο τεκμήριο της Αθότητα, αλλά και στην αρχή της αναλογικότητας των ποινών και της δικής δίκης. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε στενή επαφή με τοπικές ενώσεις όπως ομάδες πολιτών, όπως η ομάδα πολιτών που παρέχει στήριξη σε γυναίκες ε, στην δίκη τους. Με το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στηρίζουμε επίσης την παροχή νομικής αρρωγής ε, σε ε, Γυναίκε οι οποίε βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Το γεγονό ότι δεν υπάρχουν αρκετέ τέτοιε υπηρεσίε στο Ελσαλβαδόρ επίση είναι ένα εμπόδιο για να αντιμετωπιστεί το θέμα στις περιπτώσει αποβολή. και βέβαια εμποδίζει και τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα. Ο σεβασμό και η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι βασικό θέμα στη συζήτηση μας με το Ελσαλβαδόρ και αλλού. Η ολοκληρωτική απαγόρευση των εκτρώσεων που αναφέρεται στο Σύνταγμα και την νομοθεσία του Ελσαλαδόρ είναι ανησυχητική, ειδικά όταν κινδυνεύει η ζωή γυναικών και κοριτσιών ή στις περιπτώσεις βιασμού. Οι ολοκληρωτικές απαγορεύσεις είναι επίσης πρόβλημα και σε πολλές άλλες χώρες στη Λατινική Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φύγει ε, αυτό το ζήτημα στο υψηλότερο επίπεδο στο Ελσαλβαδόρ και ζητάει από την κυβέρνηση να βελτιώσει συνολικά την κατάσταση των γυναικών. Μεταξύ των άλλων πρωτοβουλειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στήριξη στο πρόγραμμα Σουηδάδ Μουχέρες, το οποίο έχει δημιουργήσει το κράτος και έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στο να έχουν πρόσβαση σε, υγείας, σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας οι γυναίκες, αλλά και στο να αντιμετωπίσει την βία με βάση το φύλλο και να ενδυναμώσει τις γυναίκες. Ενθαρρύνουμε το Ελσαλβαδόρ και τις άλλες ε, χώρες που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς αυτήν την ε, κατεύθυνση και είμαστε στην διάθεσή τους για κάθε βοήθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα έχουμε το κοινό σχέδιο ψηφίσματος. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 η ώρα και ολοκληρώθηκε η συζήτηση.